Καλημέρα σας. Να ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες παρακαλούμε. Ελπίζω να φέρατε τις κάρτες σας. ready. Έτοιμοι όλοι, κυρίες και κύριοι. Would you please take your seats? Καθίστε σας παρακαλώ. So the first, uh... Πρώτη ψηφοφορία. Έκθεση Μπέλετ, πρόταση κανονισμού για την εσωτερική αγορά, για τον ηλεκτρισμό, αναδιατύπωση, διαδικασία συναπόφασης. Τροπολογία 87 υπέρ, κατά έλεγχος. Άρχεται η συγχωρία. Πέρασε. της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 90 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 92 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 101 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. 101 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 105 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 105. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται. 106-107 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται. 108 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 109 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 11 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 110 υπέρ, κατά εποχές εγκρίνεται 111 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 111 της ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 112 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 113 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 115-116 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 143 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 146 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 148 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 149 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 150 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 224 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 225 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 226 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 227 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος. 227 έλεγχος. Δίκαιο έχετε. Μικρή διαφορά. Πέρας εγκρίνεται. 228 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 229 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 230 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 257 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 217 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 271 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η προηγούμενη ήταν 270, με συγχωρείτε. Συμβαστική 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 284 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 283 υπέρ, κατά, αποχές έλεγχος για τη 283 άρχεται πέρας απορρίπτεται 285 τι συμβαίνει Μάργαρετ 285 λοιπόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 318 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 319 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 320 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 322 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3.23 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 3.23. Πέρας. Απορρίπτεται. 3.24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Οριζόντια τροπολογία 329. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 34. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 325, 326 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 327 υπέρ. Κατά Α, ταυτόσημα. Έκανα λάθος σελίδα. 3.30. Ψηφίζουμε. 3.33 και 3.34 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 35 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 338, 39, 40 και το καθεξής. Μεγάλο κομμάτι, πολλές. Δεν διαβάζω όλους τους αριθμούς. Βλέπετε τη λίστα. Ποιος είναι υπέρ όλων αυτών μαζί. Κατά αποχές εγκρίνονται. Προχωράμε. 365 υπέρ, κατά, έλεγχος για την 365. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 36 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 37 υπέρ, κατά, Ψηφίσαμε τη 36, εγκρίθηκε. Πάμε στην 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε μια ομάδα από την 368 μέχρι την 371 υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος για, αυτό, για αυτές τις τροπολογίες. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνονται. 3.72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3.73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άλλη μια ομάδα τροπολογιών και στη 40 έχουμε προφορική τροπολογία Υπάρχει αντίρρηση όσον αφορά την προφορική τροπολογία. Όχι. Ψηφίζουμε με την προφορική τροπολογία όλη αυτή την ομάδα τροπολογιών, ξεκινώντα από τροπολογία 38 μέχρι τη 42. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 374 υπέρ κατά αποχές απόχέσ για τη 374. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Και κάποιος δεν ψήφισε. Κάποιος δεν ψήφισε. 3.75 υπέρ. Κατά έλεγχος για την 3.75. Άρχεται η ψηφοφορία. Τώρα ψήφισαν όλοι εγκρίνεται. Δεν είναι τόσο μικρή διαφορά όπως με την προηγούμενη ψηφοφορία. Λοιπόν, νέα ομάδα τροπολογιών 376 μέχρι 378 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 44. Όχι. Καταπίπτει αυτή. «3.79 υπέρ» κατά αποχές απορρίπτεται 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 382 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 382 άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 383 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 384 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 385 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 387 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 388 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 389 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μια ομάδα 390 μέχρι 392 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 48 έλεγχος για την ομάδα των τροπολογιών. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνονται. 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 394 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 397 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 50 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 54 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 421 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 422 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 423 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 424 υπέρ, κατά αποχές έλεγχος για την 424. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 425 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 426 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για 426 άρχεται η συμφορία λέει πρόεδρος πέρας εγκρίνεται 427 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για 427 άρχεται Πέρας. Α, απολύτωται. 428 και 429 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 430 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 431. Έλεγχος 430. Άρχεται. Για την 430 έλεγχος. Πέρας. Απορρίπτεται. 431. Υπέρ παρακαλώ. 431. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 432. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 433. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 434. Υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος για την 434 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 435 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 436 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 437 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 438 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 439 και 440 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 59 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται ε, εγκρίνεται συγγνώμη, 60 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 8 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 64 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 65 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 66, 67 υπέρ, 67 υπέρ, 67 δεν φαίνεται εδώ ότι καταπίπτει. Λοιπόν, 67 υπέρ παρακαλώ. Εγκρίνεται. 68 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 69 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 70 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 71 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 73 και 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 76 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 76 πέρας εγκρίνεται 77 υπέρ κατά κατά παρακαλώ 77 εγκρίνεται έλεγχος λοιπόν για την 77 άρχεται πέρας εγκρίνεται τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές Ποιος είναι υπέρ ξανά, οι δύο, εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 80 υπέρ, κατά αποχές, έλεγχος για την 80, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας απορρίπτεται. 81 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 84 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 85 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 86 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία, τελική. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Μου λέγουν ότι είπα συμβαστική 8 απορρίπτεται αλλά εγκρίνεται. Διορθώνω αυτό. Πάμε. σε άλλη έκθεση. POTS, Κοινή κανόνε για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αναδιατύπωση. Συμβαστική 8 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ, κατά έλεγχος. Συμβαστική 1. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 108 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 113 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 123 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά αποχές έλεγχος για τη συμβαστική 2. Υπάρχει ένα μέλος παραπάνω του ΕΛΚ. Παρακαλώ να βγάλετε μια κάρτα από το ΕΛΚ. Είναι ένας παραπάνω από το ΕΛΚ. Καλώς, τώρα είμαστε εντάξει. Πέρας. Απορρίπτεται λοιπόν. Συ, συμβαστική 2 απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τις τροπολογίες. 124 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 125 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 129 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 126 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 127 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 128 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 130 υπέρ κατά έλεγχος 130 έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 132 α όχι καταπίπτει καταπίπτει 134-135 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 136 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 137 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 138 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 139 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 140 υπέρ κατά υπέρ παρακαλώ. 140 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 141 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 142 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ κατά Αποχές έλεγχος η συμβαστική 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 144 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την 145. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 100. Έλεγχος για την 145. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Τυχερή ήμουνα. Απορρίπτεται. 146 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται.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 αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 153 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 154 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 155 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 156 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 157 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 158 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 159 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 160 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 164 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 200 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 201 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 202 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για τη 15. Δεν είδα ξεκάθαρα τα χέρια. Πέρας. Εγκρίνεται. 203 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 206 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κάποια διατύπωση ψηφίζουμε. Για τη 205. Υπέρ της 205. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 204 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 209 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 207 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 208 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 210 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 211 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ κατά έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. Εγκρίνεται. 212 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 213 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 214 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 215 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 216 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 217 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 218 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 219 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 17 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται μαζί 220 221 υπέρ κατά αποχές κατά μάλλον συγγνώμη 221 υπέρ εγκρίνεται 222 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 233 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 234 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 235 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 18 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 19 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 236 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 20 υπέρ, κατά Έλεγχος για την 20. Πέρας. Εγκρίνεται. 2.37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 238 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 263 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 277 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 278 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 279 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 280 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 281 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 282 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 283 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 284 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 289 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 290 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτονται 91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 92 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 93 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 94 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 298 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 299 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 300 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 301 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 302 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 303 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 304 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 306 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 305 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 307 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 308 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 310 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 311 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 309 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 26 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 27 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 28 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 29 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 30 υπέρ κατά έλεγχος για την 30 άρχεται πέρας εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τοπολογία 1 υπέρ. Κατά Αποχέ. εγκρίνεται. 36 υπέρ. Κατά Αποχέ. απορρίπτεται. 37 υπέρ. Κατά Αποχέ. απορρίπτεται. 38 υπέρ. Κατά Αποχέ. εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά Αποχέ. απορρίπτεται. 40 υπέρ κατά αποχέ απορρίπτεται, 42 υπέρ κατά αποχέ απορρίπτεται, 41 υπέρ κα, κατά αποχέ εγκρίνεται. 43. Μάλλον 45 λοιπόν. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτωται 52 υπέρ κατά κατά κατά ποιος είναι κατά 52 ωραία εγκρίνεται 53 υπέρ έλεγχος για την 52 άρχεται και τώρα τελείωσε και εγκρίνεται και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 αποχές απορρίπτεται και αυτή. 61 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 62 υπέρ. Κατά παρακαλώ επαλήθευση. 62. Α, εγκρίνεται εν τέλει. Ε, 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 65 υπέρ κατά. Επαλήθευση παρακαλώ. 65. Αρχίζει η ψήφος. Πέρας. Εγκρίνεται. 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 78 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 79 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 80 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 81 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 82 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 83 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 84 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 85 υπέρ,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 κατά αποχές εγκρίνεται αυτή. 99 επέρ. κατά. Επαλήθευση παρακαλώ. 99. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται πράγματι. Ήταν σφάλμα λέτε. Γι' αυτό είπα να επαληθεύσουμε. Γιατί είχα μια ένδειξη σχετική, αλλά εγκρίνεται πάντως. Τώρα, τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονική. Τέλος, εγκρίνεται και συγχαρητήρια. Ψηφίζουμε τώρα τον ρόλο των ε, περιφερειών για την εφαρμογή και των αστικών κέντρων για την, για την ε, εφαρμογή της COP21 του κυρίου Παρνιό για τις τροπολογίες 71 και 16 έχουν αποσυρθεί. Ψηφίζουμε την συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται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 παρακαλώ η κατά. Εγκρίνεται εν τέλει. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ Τι είπατε, λέει και η πρόεδρος. Όχι, τίποτα, εντάξει. Ε, 18. Νομίζουμε ότι κάποιος ζητεί επαλήθευση. Καλά. Ας ε, επιληθεύσουμε την 17. Τώρα τέλειωσε η ψηφοφορία και απορρίπτεται όπως βλέπετε στις όθανες. 18 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται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 κατά αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 60 70, 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 71 υπέρ κατά αποχές Α, πρώτα κατά. Ποιοι είναι κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 82 υπέρ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 Εγκρίνεται και αυτή. 91 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 92 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 93 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 94 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 95 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 96 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση.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 Επαλήθευση παρακαλώ, 111. Αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. 112 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 113 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 114 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 115 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 116 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 117 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 118 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 119 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 120 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία με ηλεκτρονική ψηφοφορία αρχίζει Εγκρίνεται λοιπόν, όπως βλέπετε, σας ευχαριστώ πολύ. Όμως, έχουμε ακόμα τις ανακοινώσεις της Προέδρου. Θα αρχίσω να σας ομιλώ καθώς αποχωρείτε, αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι πρέπει να ε, είμαστε τυπικά. Ήταν η διάσκεψη, έχουμε μάλλον διάσκεψη υψηλό επίπεδο για την Αφρική στις 21 Νοεμβρίου, αύριο λέει η Πρόεδρος, έχουμε και από δημόσιους φορείς και από ιδιωτικού φορείς συμμετοχή σε υψηλό επίπεδο, αρχίζει στις 2 το απόγευμα και πάει μέχρι στις 8 το βράδυ. Μία από τις τόγγυλες τράπεζες θα ασχολείται με την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, κάτι το οποίο νομίζω μας ενδιαφέρει Έχουμε επίσης ε, και την ομάδα εργασίας ε, που οργανώνεται από την ομάδα την οποία συμπροεδρεύουν οι Καμπεζόν και ο Πέτερλε και από τις 10 μέχρι τις 12 αύριο προσκαλούνται όλα τα μέλη να πάρουν μέρος. Έχετε και μία έκθεση από την ε, αποστολή στην διάσκεψη για τους ωκεανούς το μήνα Ιούνιο των Ηνωμένων Εθνών σε σχέση με τις διοργανικές διαπραγματεύσεις τώρα που εξελίσσονται για το EGS έχουμε την προσωρινή συμφωνία στα πλαίσια του έκτου τριμερούς διαλόγου στην τέταρτη φάση του συστήματος εμπορίας εκπομπών. Από θεματικό σταθερότητας, γραμμική μείωση 2,2, μείωση των πληστηριασμών έτσι ώστε να αποφύγουμε την εφαρμογή του παράγοντα του διορθωτικού εξαίρεση της ομαδικής θέρμανσης. 02 1,6%. 50 εκατομμύρια για το Ταμείο Καινοτομίας όχι υποστήριξη για τα Cohen Generation. With a GDP per capita below 30% of the EU average and possible support for just transition in carbon Στα θέματα συμπαραγωγής ενέργειας, εκεί δεν θα υπάρξει υποστήριξη. 0,5% αύξηση μετά από την εφαρμογή του γραμμικού ε, παράγοντα διόρθωσης κριτήρια τα οποία επίσης ε, εφαρμόζονται μετά από την ε, εξαίρεση του άρθρου σε Μια πράξη κατ' εξουσιοδότηση επίσης από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την οποία θα πρέπει να εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Να πω ότι στις 2.30 μόνο σήμερα το απόγευμα Έχουμε την υπεύθυνη διευθύντρια ε, του Παγκόσμιου Οργανικού Υγείας για την Αφρική και σας παρακαλώ να είστε εδώ στις 2.30 για την παρουσίαση αυτή. Σας ευχαριστώ.